is an independent... Είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος ο κύριος Γιγέρμο Φαρίνας και πολιτικός αντιφρονών και ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του την ίδια ως μέσο πίεσης για να αλλάξει η κατάσταση στην Κούβα μέχρι και σε απεργία πείνας κατέληξε για να βοηθήσει όλους εκείνους που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία προσωπικά να του απονείμω το Δεκέμβριο εδώ στο Στρασβούργο το βραβείο Σαχάροφ. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και για όλους τους κρατουμένους συνείδηση στην Κούβα. Ειλικρινά ελπίζω μαζί με τον ε, Γιγέρμο Φαρίνας είναι και οι κυρίες με τα λευκά, η Ντάμας Ντεμπλάνκο που βραβεύτηκαν το 2005. Ελπίζω να έχουν την ευκαιρία και οι κυρίες ε, εκείνες να έρθουν στο Στρασβούργο. Αυτό Πρέπει να θυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι ήταν εξαιρετικοί όλοι οι υποψήφοι από πλευράς ε, της αντίληψης που έχουμε εμείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το πώς αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο και όλους τους συγχαίρουμε. Αλλά έπρεπε να κάνουμε μία επιλογή, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι παντού στον κόσμο έχουμε πολλούς βραβευτέντες και τους υποστηρίζουμε όλους. Ας το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα συνάδελφοι. Το πρώτο θέμα διαδικαστικό έχετε παρακαλώ. Η κυρία Βερζιά. Εγώ θέλω να αναφερθώ στον κανονισμό. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον, τον οποίο αποφασίστηκε το βραβείο Ζαχάρφ είναι σκανδαλώδης διότι η πολιτική θεώρηση υπερισχύει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η τρίτη φορά μετά από την ίδρυση, από τη θέσπιση του βραβείου Ζαχάρο. Εγώ πάντοτε πάλεψα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όποια και να, να είναι αυτά αλλά εδώ και 20 χρόνια που υπάρχει το βραβείο Ζαχάροφ τρεις φορές έχει δοθεί σε κουβανούς. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε και αυτό υποβαθμίζει το βραβείο Ζαχάροφ. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ το βραβείο Ζαχάροφ να μην αποφασίζεται στη διάσκεψη των Προέδρων αλλά συνολικά από όλους τους βουλευτές Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, με ενημερώνουν ότι έγινε πολύ εκτενή συζήτηση και σε μεγάλο βάθος.